καλό απόγευμα. Θα μάθετε κι άλλες λέξεις σήμερα το απόγευμα. Σας ξαναλέω καλημέρα σας στα Ιταλικά. Apriamo la nostra riunione della... Αρχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να πληροφορήσω τους συναδέλφους ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω του ίντερνετ, web stream. Έτσι ε, να προσπαθούμε όλοι να φαινόμαστε πιο όμορφοι και να είμαστε πιο καλοί σε αυτά που λέμε. Ε, παρακαλώ να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Περνάω στο σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών. Συνεδριάσεις 20 και 22 Ιανουαρίου. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε αντίθετα σχόλια. Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης προθεσμία για σχόλια. Σημείο 3. Έχω το προνόμιο να μπορώ να καλωσορίσω τον Υπουργό Πέτρε Μπέγκλ, Υπουργό Μεταφορών της Τσεχίας, η οποία έχει και την Προεδρία του Συμβουλίου Μεταφορών. Και θα συνεργαστούμε με την Προεδρία όλο αυτό το εξάμεινο. Όπως ξέρετε, από τις ε, από την ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε θα είναι μια ευκαιρία για μια πρώτη συνάντηση για να οργανώσουμε τις εργασίες μας για όλο το εξάμεινο. Δεν θα φάω άλλο χρόνο, όπως ήθιστε. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον Υπουργό κύριο Μπέντο να μας παρουσιάσει τις απόψεις του. Και σας διαβεβαιώνω κύριε Προεδρεύοντα, οι συνάδελφοι με ευχαρίστηση θα αντιδράσουν, θα σχολιάσουν, έτσι ώστε η δουλειά μας να είναι όσο πιο αποτελεσματική γίνεται. Έχετε το λόγο. Hezký dobrý den, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να σας συναντήσω σήμερα και να σας ε, ε, παρουσιάσω τις προτεραιότητες της τσεχικής προεδρίας στον τομέα των μεταφορών στην ε, αρμόδια επιτροπή. Είμαι νέος υπουργός μεταφορών και οι μεταφορές για τη χώρα μας ήταν πάρα πολύ σημαντικές πάντοτε διότι όλες οι μεταφορές περνούσαν από τη χώρα μας. Μετά από την ε, πτώση της, ε, του σιδηρού παραπετάσματος και την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση επανακτήσαμε την ε, θέση μας στον χώρο των μεταφορών και είμαι υπουργό της Βοημίας που ασχολείται με το θέμα αυτό. Και είμαστε εξαιρετικοί σε ορισμένα θέματα, διότι ο αριθμός των επιβατών στα δημόσια μέσα στην Πράγα είναι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και έχουμε πάρα πολύ στενό δίκτυο τουριστικών περιπάτων στη χώρα μας. Θέλω να είμαι θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν ε, συμφωνώ βέβαια με τον κύριο Σαρκοζή να μεταφερθεί η αυτοκινητοβιομηχανία γαλλικών συμφερόντων από την Τσεχία ή στη Γαλλία και ελπίζω θα αλλάξει γνώμη. Αλλά ευχαρίστω θα συνεργαστώ μαζί σας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους στον τομέα των μεταφορών θα προσπαθήσουμε να ε, καλύψουμε ως το δυνατόν περισσότερους τομείς μεταφορών κατά την Προεδρία μας ε, και έχουμε τρεις βασικούς στόχους την αηφορία και την ανταγωνιστικότητα των μεταφορών, την ασφάλεια των μέσων μεταφοράς και την ε, ανάπτυξη εξύπνων συστημάτων μεταφοράς. Ένα άλλο βασικό θέμα είναι η οργάνωση του χρόνου εργασίας οι οποίοι ε, κινούνται ε, για, την, ε, για επαγγελματικούς λόγους διότι έχουμε μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια και υπάρχει μία ασαφής περιοχή μεταξύ των επαγγελματιών οδηγών και των ήμι επαγγελματικών οδηγών γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να διορθώσει ολοκληρωθώ στην κατάσταση μέχρι το 2015 και έχουμε ξεκινήσει υπό Προεδρία της Τσεχίας να καταρτίζουμε αυτή την νομοθεσία και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Τώρα λίγα λόγια σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σήμα, την Eurovignette διότι παρόλο που το θέμα είναι περίπλοκο, όπως ξέρετε υπάρχει στόχος ε, να εφαρμόσουμε στις μεταφορές την αρχή ότι ο ρηπαντής πληρώνει και πρέπει να είναι λειτουργικό το σύστημα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί ε, να ε, διεκπαιρεώσει εκ των έσω αυτή, αυτό το θέμα, άρα θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα είναι δυνατόν να προστατέσουμε το περιβάλλον και το δικό σύστημα και πώς θα βρεθεί ένα σύστημα διοδίων που θα επιτρέψει στους μεταφορές, ε, μεταφορείς να χρησιμοποιούν ε, οχήματα πιο φιλικά στο περιβάλλον και ε, όχι όλοι τους ίδιους δρόμους. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν αρχές οι οποίες είναι σωστές, πρέπει όμως να είμαστε και Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ περίπλοκο το θέμα αυτό, γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε να ισοσκελίσουμε την κατάσταση και να καταλήξουμε σε μία συμφωνία. Θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το θέμα αυτό κατά την Τσεχική Προεδρία, η οποία ούτως ή άλλως θεωρεί ότι μία από τις προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, να ανταποκριθεί συγκεκριμένα στις ανάγκες των πολιτών. Γι' αυτό και έχω δύο προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους όταν χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς και γι' αυτό χρειαζόμαστε να υπάρχουν κοινά αποδεκτά δικαιώματα. Έχουν ε, υιοθετηθεί ε, νομοθετήματα ζητήματα σχετικά με τις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και έχουμε επικεντρωθεί στην ασφάλεια των θαλασσών. Προσφάτως συμφωνήσαμε με το Κοινοβούλιο για την ευθύνη, ε, την αστική ευθύνη των ε, ε, εφοπλιστών σε περίπτωση ατυχημάτων και θα πρέπει να στελεχώσουμε το οικοδόμημα που έχουμε δημιουργήσει για τους πολίτες σε αυτό το σημείο θα ασχοληθούμε ιδίω με τρει τομεί επιπλέον, με τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, την ε, απώλεια αποσκευών ή την απώλεια ζωής ή τα ατυχήματα και τις ε, και ε, ε, τις αποζημιώσεις. Η δεύτερη πρόταση αναφέρεται στους επιβάτες και των θαλασσίων μεταφορών και των ποταμίων μεταφορών και ε, θέλει να καλύψει όλους τους επιβάτες, να τους ενημερώσει για τα ε, δικαιώματά τους και να διεκπεραιώνει τα παράπονα. Ελπίζουμε δε ότι κατά το επόμενο εξάμεινο θα μπορέσουμε στον τομέα αυτό να έχουμε προχωρήσει επαρκώς και αναφέροντας τα δικαιώματα των επιβατών των θαλασσίων μεταφορικών μέσων έρχομαι να μιλήσω και για τις θαλάσσιες μεταφορές διότι η Τσεχία είναι μία χώρα στο εσωτερικό έχουμε περιορισμένες δυνατότητες είμαστε όμως ευγνώμονες στην προσεχή Σουηδική Προεδρία με την οποία συνεργαζόμαστε στενά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οθετήσει ζητήσει μια ανακοίνωση σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους όσον αφορά τις ε, θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 που αναφέρονται τα βασικά σημεία και καταρτίζονται οι προτεραιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής για το συντονισμό της ναυτιλιακής πολιτικής. Υπήρχε και μία ανακοίνωση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Χωρίς Σύνορα που είναι ένα από τα θέματα που διεκπαιρώνει η Τσεχική Προεδρία, δηλαδή να καταργήσουμε ε, τους φραγμούς. Επίσης θα ασχοληθούμε και με την αεροπορία, διότι όπως ξέρετε τον περασμένο Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ορισμένα μέτρα, ένα πακέτο σχετικά με την ε, Ευρώπη των ενιαίων ουρανών και είναι κάτι το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε από το 2004 για να υπάρχει υπάρχει ένα ενιαίο οργανωμένο σύστημα ε, των ε, ε, ελέγχων του αεροπορικού χρόνου, να εξυγχρονίσουμε τον στόλο των αεροπλάνων και στον εξοπλισμό και συγχρόνως να δημιουργήσουμε τις αναγκαίες περιποθέσεις για τις σύγχρονες αεροπορικές μεταφορές. Όλα αυτά έχουν σχέση με τις δυνατότητες και το αβάρι επί του συστήματος. Είναι πολύ σημαντικά. Ελπίζουμε ότι θα εμποδίσουμε το κατακαιρματισμό στις αεροπορικές μεταφορές για να μπορέσουμε να υποφεληθούμε από όλες τις δυνατότητες του συστήματος και κατά αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουμε και την ασφάλεια ασφάλεια και να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Η Τσεχική Προεδρία θα συνεχίσει το έργο της Γαλλικής Προεδρίας στο θέμα αυτό και στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου επιτύχαμε μια γενική συμφωνία για τα τεχνικά θέματα του κανονισμού για τους ενιαίους ε, ουρανούς, το single skies όπως λέγεται και θα θέλαμε να επιτύχουμε με το Κοινοβούλιο μία συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ήδη έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους εισηγητές Μαριάντζελα Μαντνέσκου και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό εντός της θητείας του παρόντος Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο των Υπουργών θα ήθελε ε, να μπορέσει να υιοθετήσει και το πρόγραμμα των ε, θαλασσίων μεταφορών. Επίσης έχουμε ε, προτείνει μία αναμόρφωση του δευτέρου προγράμματος Μάρκο Πόλο το οποίο θα βελτιώσει την, τις μεταφορές ως προς, τις, ως προς πιο φιλικές για το περιγάλλον και έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την μετακίνηση προς άλλων ειδών μεταφορές ότι το Μαρκοπόλο δεν καλύπτει όλες τις απαιτήσει, άρα έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση με μέχρι 525 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο ένα μικρό ποσοστό της χρηματοδοτήσεως αυτής Άρα θα πρέπει να το προσαρμόσουμε για να είναι πιο αποτελεσματικό, να ε, προσφέρει ορισμένα οικονομικά κίνητρα, ιδίω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διότι θεωρούμε ότι αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικό και θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις και να επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις. Έχουμε ήδη επαφή με με τον εισηγητή κύριο Στόκμαν. Και τώρα θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το μέλλον του ε, διευρωπαϊκού δικτύου TNT διότι ε, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης είναι απαραίτητο να εξετάσουμε την υποδομή των μεταφορών να υποκινήσουμε δημιουργία θέσεων εργασίας, ανάπτυξη και ορισμένα κράτη έχουν τέτοιες ε, προτάσεις και προσπαθούμε συγχρόνως να βρούμε μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για συστήματα συστήματα τα οποία θα βελτιώσουν την απασχόληση και θα μπορέσουν να συνδέσουν διάφορες περιοχές, νέες δηλαδή συνδέσεις μεταξύ της Βαλτικής και της Αδηρετικής. Είναι ένας από τους στόχους μας. Και μέχρι το Δεκέμβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μελετήσει τις προτάσεις που θα μπορούσαν να χρηματοδοτικούν. Υπάρχει και ένα, ε, ε, ένα επιπλέον ε, πρόγραμμα ε, για τα ε, δίκτυα και θέλουμε να μπορέσουμε έτσι να ενισχύσουμε και τις οικονομίες των κρατών μελών. Οπότε με, στα πρέσια αυτών των τέντι θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τις μεταφορές και τέλος θέλουμε να ολοκληρώσουμε τις αποφάσεις όσον αφορά το πακέτο οδικών μεταφορών και να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την νέα οδηγία για το Ευρωπαϊκό Σήμα. Όσον αφορά το, τις οδικές μεταφορές, ελπίζω ότι όλοι θα είναι επαρκώς ευέλικτοι για να, να καταλήξουμε σε μία συμφωνία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουμε την κατάσταση των επιχειρήσεων, να μειώσουμε το διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις επιχειρήσεις αλλά και για τα θεσμικά όργανα και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα συγχρόνως δεσμεύοντας όλους τους χρήστες να καλύψουν τις προϋποθέσεις ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο συμμερίζεται αυτές τις απόψεις στα πλαίσια της ανοιχτή αγοράς και γι' αυτό ελπίζω ότι θα υπάρξει ε, ε, μνήα των διαφορετικών οικονομικών καταστάσεων των διαφόρων χωρών κατά τρόπον ώστε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό και να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία αυτή Γι' αυτό ο, συνεργαζόμαστε με την κυρία Σίλβια Τικάου και τον κύριο Άντριαν Γκρός. Προτού ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για τα μελλοντικά μας σχέδια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την προσοχή σας και την υπομονή σας δεν θα έχουμε έξι μήνες για να συνεργαστούμε μαζί. Θα πρέπει όλα να έχουν διεκπαιρεωθεί σε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε λιγότερο χρόνο. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να καταρτήσουν προτεραιότητες, να δούμε ποιες μπορούν να διεκπαιρεωθούν προτού ολοκληρωθεί η θητεία αυτού του Κοινοβουλίου, να συνεργαστούμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και πιο στενά και δεν θα αφήσουμε ε, την ε, τσεχική ολιγορία να υπερισχύσει αλλά θα προσπαθήσουμε γρήγορα να καταλήξουμε ε, σε ρεαλιστικές λύσεις και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Πιστεύω δε ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες για να συζητήσουμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα των μεταφορών στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Eh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Υπουργό. Βγαίνετε με την τελευταία πρόσκλησή σας από κοινού να ορίσουμε μια αποτελεσματική σε διάταξη για το τελευταίο αυτό και για μας τελευταίο εξάμεινο. για να δούμε στην πράξη πώς θα δοκιμάζεται η βούλησή μας να βρούμε καλές λειτουργικές λύσεις που ανταποκρίνονται προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που εκπροσωπούμε. Αρχίζουμε έναν πρώτο γύρο παρεμβάσεων, συντονιστές. Ο κύριος Γιαζεμπόφσκι πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την εξαιρετική εισαγωγή. Σας ευχόμαστε καλή η υπηρεσία, θα συνεργαστούμε ευχαρίστως και πρέπει να σας πω ότι τα τσεχικά αυτοκίνητα είναι εξαιρετικά και τεχνολογικά αλλά και από πλευράς χρήσεως και ε, αν βλέπουμε πώς έχουν ε, ε, κατασκευαστεί τα τσεχικά Audi είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στο τι μένει ακόμη να διεκπαιρεωθεί. Και σαν πολιτική ομάδα έχουμε δύο θέματα τα οποία μας απασχολούν πολύ και τα οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε πριν αποχωρήσουμε. Το, το ε, πακέτο Gross για την μεταφορά μέσω οχημάτων ε, και νομίζω ότι συζητούν μαζί σας, δηλαδή θέλουμε και ασφάλεια αλλά και ρύθμιση ε, μέσω του κλάδου για ε, τους, την ασφάλεια των επιβατών. Υπάρχει και ο χρόνος εγγυήσεως και όλα αυτά πρέπει να λάβουν υπόψη και την αστική τάξη η οποία αποτελεί ε, τη γραχοκοχαλιά της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Και έχουμε επίσης και την έκθεση ε, Τικάου Εάν λοιπόν δεν καταφέρουμε να καλύψουμε αυτά τα δύο σημεία θα είναι πολύ δυσάρεστο, θα έχουμε χάσει ουσιαστικά ένα χρόνο και θα θέλαμε για λόγους κόστους, για λόγους Ε, Αν δεν έχουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, το χρειαζόμαστε ένα αλλά τα άλλα τα χρειαζόμαστε πιο πολύ και ε, θα έπρεπε περισσότερο να μας απασχολήσει το θέμα του Ευρωπαϊκού Γραφείου των, ε, ε, της ασφαλείας των αερομεταφορών και η έκθεση του θα έπρεπε να διεκπεριωθεί. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μας. Ε, αυτό που δεν είναι προτεραιότητα για τη δικιά μου πολιτική ομάδα είναι το Ευρωπαϊκό Σήμα και αυτό για δύο λόγους. Βεβαίως κάνουμε εδώ μια πολιτική συζήτηση και παρουσιάζουμε πολιτικά επιχειρήματα. Για δύο λόγους λοιπόν, διότι αν δείτε ε, ποια είναι η κατάσταση του μετακομιστικού εμπορίου ε, στην Ευρώπη, υπάρχει μεγάλη δυσκολία, οι εταιρείες διώχνουν προσωπικό, και εφόσον ούτως ή άλλως θα χρειαστεί και έχει προβλεφτεί μία αναθεώρηση θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά πώς θα προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει καμία βία διότι η εφαρμογή ε, ε, του μέτρου αυτού ήδη έχει προβλεφθεί. Άρα δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι σωστό διότι οι οδικές μεταφορές είναι βασικό θέμα και αν δώσουμε λανθασμένο σήμα θα αντιμετωπίσουμε δυσκολία. Προ προς σοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους έχω να πω ότι οι συμφορήσεις οι οδικές δεν είναι δυνατές αλλά γι' αυτά ευθύνονται τα κράτη διότι δεν μπορέσανε να βελτιώσουν το δικό τους σύστημα και εφόσον ε, δεν υπάρχει καλό δικό σύστημα δεν υπάρχει λόγο μεταφορέας να πληρώνει περισσότερο για τα λάθη των ε, εθνικών διοικήσεων. Ασχέτως των απόψεων θα το συζητήσουμε και το Συμβούλιο θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά πώς θα προχωρήσει. Γι' αυτό για λόγους ε, περιβάλλοντος δεν υπάρχει λόγος αυτό να διεκπαιρεωθεί γρήγορα. Κάτι προβλέπεται για ε, μια περαιτέρω ημερομηνία και είναι καλύτερα πιο σημαντικό εδώ να μην βιαστούμε αλλά όσον αφορά τις δύσκολες καταστάσεις των μεταφορικών επιχειρήσεων να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στη σωστή απόφαση. Και τελευταία παρατήρηση θέλουμε να διεκπαιρεώσουμε και τα δικαιώματα των επιβατών αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όταν κάνουμε κάτι πρέπει να σκεφτούμε και τις δύο πλευρές, διότι η δικιά μας ε, ε, πολιτική ομάδα ε, ζήτησε να καλυφθούν τα δικαιώματα των επιβατών αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα λεωφορεία και τα φέριμποτ και τις κρουαζιέρες. Ο συνάδελφος Αλμπερτίνη έκανε μια θαυμάσια έκθεση ε, κοιτάζουμε όλα αυτά τα δικαιώματα, αλλά χρειάζεται να είναι ισοσχελισμένα, ισορροπημένα και ε, να διεκπαιρεώσουμε ό,τι είναι έτοιμο και ό,τι άλλο χρειάζεται περαιτέρω σκέψη, να το αφήσουμε να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Σας ευχαριστώ. Thank you, President. I thank the President in Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριο κύριο Σίμψον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Προεδρεύοντα για την εισαγωγή του, γιατί μεταξύ άλλων ε, κατάφερε να βγάλει τη θέση του Γιώργου Γιαρζεμπόφσκη σχετικά με το ευρωπαϊκό σήμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για τον ε, ευρωπαϊκό ουρανό, ενιαίο ουρανό, χρειαζόμαστε αυτό και εκείνο για να βοηθήσουμε το περιβάλλον, λέει. Όταν ερχόμαστε στο ευρωσήμα τελών κυκλοφορία δεν το θέλουμε. Οι πιο μεγάλοι ρηπαίνοντε είναι τα φορτηγά. Δεν το θέλουμε όμω αυτό. Υπάρχει μια ανακολουθία εδώ. Ξέρω, κύριε Προεδρεύοντα, ότι μάλλον πρώτη φορά άρχισε το όσοι από εμά είμαστε εδώ εδώ και χρόνια και έχω συνεργαστεί με τον ε, Γιώργο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τέτοιου είδους ανακολουθίες δεν με ξαφνιάζουν. Σε όσα μας είπατε, θέλω να τα περισσότερα τα δέχομαι. Ένα μόνο που θέλω να πω είναι ότι είπατε πολλά είναι σαν να πάτε να ψωνίσετε σε ένα σούπερ μάρκετ με ένα κατάλογο των πραγμάτων που θέλετε να αγοράσετε, εδώ προκειμένου που θέλετε να κάνετε. Αν τα καταφέρνετε να τα κάνετε όλα αυτά που είπατε, θα ήταν μνημειώδης η προεδρία σας και θα τη θυμόμασταν για πάρα πολλά χρόνια. Απ' την άλλη μεριά καταλαβαίνω την ανάγκη να κινηθούμε, να προχωρήσουμε σε ορισμένα θέματα θέλετε να κλείσει το, θετικά το θέμα της, του Ευρωπαϊκού Σήματος και των Ενιαίων Ουρανών. Ας έρθουμε όμως στα δικαιώματα των επιβατών. Ε, συγγνώμη, να είμαστε λίγο κοινικοί για τα δικαιώματα των επιβατών, γιατί πιστεύουμε ότι είχαμε μια καλή νομοθεσία για επιβάτες της αεροπορίας. Αυτό που είδαμε όμως, οι εταιρείε κατάφεραν να βρουν παράθυρα στο νόμο λόγω να μην πληρώνουν ε, αποζημιώσεις στους επιβάτες που δεν θα μπορούσε αυτό να το φανταστεί κανένας αυτά που γίνεται. Το μόνο λοιπόν που θέλω να πω και να ζητήσω αν μιλάμε για δικαιώματα των επιβατών ο νόμος πρέπει να είναι απολύτως στεγανός να μην δίνει την ευκαιρία στις εταιρείε να υπεκφεύγουν των ευθυνών τους. Μια ευκαιρία που τους δόθηκε στις αεροπορικές εταιρείες και σε κάθε ευκαιρία την εκμεταλλεύονται αυτή τη δυνατότητα μέχρι τώρα. Γιατί δεύτερη συμφωνία, δεύτερη φάση συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Όλοι λέμε ότι συμφωνούμε, το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν αν θα συμφωνούμε εμείς με εσά, είναι ότι γίνεται από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, αν αυτοί συμφωνούν. Και όσοι από εμά παρακολουθούμε το θέμα αυτό εδώ και χρόνια, ξέρουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι από τη δική μας πλευρά του Ατλαντικού. Το πρόβλημα έγκυται βρίσκεται μάλλον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και για να δούμε τι θα κάνει η Τσεχική Προεδρία έτσι ώστε οι Αμερικάνοι να έρθουν στις διαπραγματεύσεις με λίγο πιο ανοιχτό πνεύμα. Αναφήκατε στην οδική ασφάλεια. Για το πρόγραμμα δράσης για την αστική κινητικότητα. Για την οδική ασφάλεια πρώτα-πρώτα. Το Κοινοβούλιο είναι υπέρ της ασφάλειας αυτής εδώ και χρόνια. Πιέζουμε για το θέμα αυτό. Ποιος μπλοκάρισε την πρόοδο για την οδική ασφάλεια? Τα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο μπλοκάρει, γιατί δεν θέλουν να απεμπολίσουν διάφορες εξουσίες που έχουν. Ωραία αυτά που μας λέτε για την οδική ασφάλεια. Θα σας έλεγα όμως, και το ίδιο ισχύει και για μερικά άλλα θέματα, για τη μεταφορά φορτίου με του σιδηροδρόμου κλπ. Φροντίστε να έχετε τη δική σα πλευρά συμπαγή και σύμφωνη πριν έρθετε να συζητήσετε με το Κοινοβούλιο και να ζητήσετε δική μα συμφωνία. Εμεί είμαστε η εύκολη πλευρά, Πρόεδρε. Η δύσκολη πλευρά είναι η συνάδελφοί σα, στο Συμβούλιο. Πρόγραμμα δράση αστική κινητικότητα. Ναι, θέλουμε η Κομισιόν να προχωρήσει. Μα υποσχέθηκε ότι θα προτείνει ένα τέτοιο σχέδιο. Δεν το έκανε λέει ωραία λυρικές φράσεις κλπ, δικαίωμα πρωτοβουλία κομισιών, πολύ ωραία. Ας τους δούμε να αντασκούνε τα δικαιώματα αυτά όμως. Για το πρόγραμμα δράσης για την αστική κινητικότητα, ίσως από κοινού θα μπορούσαμε να τους πιέσουμε να διορθώσουν, να επιλύσουν μάλλον τις εσωτερικές τους δυσκολίες για το πλάνο αυτό. Σε τέλος, είπατε συνεργασία. στο λίγο χρόνο που έχουμε να πετύχουμε αποτελεσματική δράση. Οι σοσιαλιστές θα συνεργαστούν, οι συγητές και όδες συγητές, εγώ συντονιστής θα συνεργαστούμε με εσά προκειμένου να το πετύχουμε στο εξάμεινο αυτό. Αλλά ξαναλέω, αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι, θα το κάνουμε με εσά, αλλά οι άλλοι συναδελφοί στο Συμβούλιο είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Βαντα. Μας ε, απαριθμίσατε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και ελπίζω θα μπορέσετε να διευθετήσετε ένα μεγάλο μέρο αυτών μέχρι το τέλο τη Προεδρία ή τουλάχιστον να κάνετε να προχωρήσουν τα πράγματα. Θα είναι μεγάλο κατόρχο, δεδομένου ότι έχετε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας και έχουμε και την προεκλογική εκστρατεία της ευρωεκλογίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτά τα οποία είπατε στην αρχή όταν μιλήσατε για την ε, αυτοκινητοβιομηχανία και όλα τα σχόλια περί αυτής. Όντως, υπάρχει κίνδυνος για την εσωτερική αγορά. Και ας μην ξεχνούμε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι μία σοβαρή εγγύηση για τον εύρυθμο τρόπο λειτουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής, εσωτερικής αγοράς. Τώρα, αυτά που έλεγε ο κύριος Γιαρζεμπόφσκι προηγουμένως, δηλαδή το ότι το Κοινοβούλιο στο περίφημο πακέτο σχετικά με το θέμα αυτό πρότεινε κάποια πράγματα θετικά. Εγώ πιστεύω ακόμη και, σε, και για την ακτοπλή. Εγώ πιστεύω ότι αντιθέτως είμαστε αρκετά περιοριστικοί σε αυτά που κάναμε. Βεβαίως δεν θα πρέπει να επανέλθουμε σε όλα αυτά τα θέματα και δεν θα πρέπει να περιορίσουμε και την, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα των μεταφορών. Θα είναι κρίμα. Και βεβαίως καταχρήσεις γίνονται. Το λέει και η έκθεση τη κυρία Δετίκα και θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε για να περιορίσουμε τις καταχρήσεις. Αλλά στην ενιαία εσωτερική αγορά θα πρέπει να είμαστε αυστηροί και σοβαροί και από τη στιγμή που κάνουμε κάτι θα πρέπει να το κάνουμε συνεκτικό τρόπο. Ένα άλλο θέμα είναι το περίφημο ευρωπαϊκό σήμα, η Εγωβινιέτ. Όπως ξέρετε, αύριο στο Κοινοβούλιο θα ψηφίσουμε την ε, έκθεση που αφορά το Ευρωπαϊκό Σήμα. Έχουν κατατεθεί διάφορες τροπολογίες από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Ε, ξέρετε που βρισκόμαστε περίπου. Και θα ήθελα να μου πείτε εσείς που βρίσκεστε στο Συμβούλιο, ποιες είναι οι θέσεις και των μεν και των δε. Διότι πολλές φήμες ακούγονται δεξιά και αριστερά και θα ήθελα ο Προεδρεύων να μας πει περί τίνος πρόκειται. Ακόμη και με, για τις οδικές μεταφορές θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις. Εγώ πιστεύω ότι τα επόμενα 20 χρόνια όχι μόνο θα πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, οδικές ε, μεταφορές και γενικότερα να βελτιώσουμε την κατάσταση, αλλά... Er το ίδιο να κάνουμε και, στις, και για τις θαλάσσιες μεταφορές. Διότι φτάσαμε στα ανώτατα όρια και θα πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα, να αλλάξουν. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα μεταξύ των μεταφορών, των τελωνίων και τι γίνεται στο Συμβούλιο σε αυτό το θέμα. Επίσης, για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Ξέρουμε ότι προβλέπεται κάτι για να μπορέσουν να εξελιχθούν οι ευρωπαϊκοί ε, σιδηρόδρομοι. Θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί το νομικό πλαίσιο, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγματα με περισσότερες λεπτομέρειες. Τι προβλέπετε για να υπάρξει πρόοδο στον τομέα αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις εκ μέρους των κρατών μελών, γιατί πρέπει να, πρέπει να λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά χρειαζόμαστε τις ιδεοδρομικές μεταφορές, το σιδηρόδρομο γενικότερο, αν θέλουμε ένα μέρος των οδικών μεταφορών να μεταφερθούν σιδηροδρόμους. Τα δικαιώματα των βιβατών επίσης είναι σημαντικό θέμα. Ξέρουμε ότι υπάρχει κάποια μικρή πρόοδος για τις θαλάσσιες μεταφορές. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε κάτι διότι όπως είπαμε και το έχω πει πολλές φορές και στην Κομισιό θα πρέπει να έχουμε μια υγιή εσωτερική αγορά. Πρέπει λοιπόν να κάνετε πολλή δουλειά. Έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας και σας ευχαριστώ για το πνεύμα στην που επιδείξατε. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και την ε, ευκαιρία να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτά ακόμη και με τις επόμενες προεδρίες. Ευχαριστώ κύριο Κράμερ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας. Επίσης ε, ελπίζουμε ότι θα συνεργαστούμε καλά το επόμενο εξάμεινο. Έχετε ακόμη ε, δύσκολα θέματα μπροστά σας όσον αφορά τους πρασίνους και τις οδικές μεταφορές. Επίσης έχουμε πει ότι η συγχρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάει κατά 60% στις οδικές μεταφορές και 40% στις ε, σιδηροδρομικές. Έχουμε προβλήματα με τις γειτονικές σας χώρες όπου δεν ε, ε, λειτουργούν ορισμένες σιδηροδρομικές αρτηρίες και ζητούν μια ενίσχυση χρηματοδοτήσεως για τους σιδηροδρόμους. Το Συμβούλιο μπλοκάρει αυτή τη δυνατότητα και αναρωτιέμαι αν εσείς θα μπορούσατε να δείτε μια διέξοδο για να μπορέσει με τη συγχρηματοδότηση να δοθεί ο σωστός προσανατολισμός ή ε, την ε, πολιτική μεταφορών. Σχετικά με το ευρωπαϊκό σήμα διαφέρουν οι απόψεις, αλλά πρόκειται για τη μείωση των προτερημάτων. Δηλαδή, οι οδικές μεταφορές είχαν εδώ και δεκαετία πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά προτερήματα, τα οποία απλούστατα υπήρχαν σε περιορισμούς για το σιδηρόδρομο και μετά τόνους για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, πολλά, ε, ε, πολλά προγράμματα αλλά όχι για να προωθηθούν οι μεταφορές από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές αλλά αντιστρόφως. Και γι' αυτό κύριε Γιαρζεμπόσχη ελπίζω ότι σε μερικές εβδομάδες που έχουμε ακόμη καιρό στη θητεία μας θα το έχετε καταλάβει. Ε, πάντοτε υπάρχουν ευκαιρίες. Επίσης οι επιβάτες με απασχολούν επίσης διότι έχουμε 50% ε, αποζημίωση για τους επιβάτες στο σιδηρόδρομο εάν υπάρχουν δύο ώρες καθυστέρηση και 25% για μία ώρα καθυστέρηση. Ξέρετε όμως ότι ορισμένα κράτη έχουν ζητήσει να μπορέσουν ε, να ε, συνεχίσουν τις εξαιρέσεις ή εσείς θα ζητήσετε το μέτρο αυτό να εφαρμοστεί γρήγορα τώρα με την έκθεση Μπισό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι εμπορευματικές μεταφορές θα πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε ορισμένους τομείς. Εγώ όμως εις την ε, έκθεση μου απέρριψα μία τέτοια λύση γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μία μεικτή διαχείριση ε, που συνδυάζει μεταφορές επιβατών και ε, ε, αγαθών. Επίσης σχετικά με το σύστημα, με τα, με τα φορτηγά της Μόντσα. Ο συνάδελφος λέει οικολογικά. Μην το πιστεύετε όμως. Ε, θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν εσείς θα επιμείνετε για να μπορέσει να ε, προωθηθεί η χρήση αυτών των φορτηγών αυτοκινήτων σε όλη την Ευρώπη. Επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε έναν ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο. Υπάρχουν σύνορα Νομίζω ότι αυτό ισχύει ακόμη και μεταξύ χωρών ή στη Βόρειο Θάλασσα και στην Βαλτική. Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να έχουμε μόνο μία εσωτερική αγορά αλλά και μία εσωτερική θάλασσα. Και ε, χρειάστηκαν 20 χρόνια για να πέσει ο τείχος του Βερολίνου αλλά νομίζω ότι θα πρέπει αυτή η πολιτιστική τάση να μπορέσει να προωθηθεί κατά τρόπον ώστε να θυμηθούμε την Προεδρία σε και τη φετινή χρονιά και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, η αναφορά σας ότι η πολιτική σας καριέρα άρχισε με την πτώση του σιδηρού παραπατάσματος, όπως ισχυριστήκατε, δεν πρόκειται να εξαγνίσει ούτε να συγκαλύψει ότι η περίοδος που διανύουμε είναι μια κρίσιμη που χαρακτηρίζεται με κρίση οικονομίας και στα 27 κράτη-μέλη και γενικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με σοβαρά οξυμένα προβλήματα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, οι μεταφορές οι οποίες είναι στρατηγική σημασίας τομής για την οικονομία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικότερα για τους λαούς των 27 κρατών μελών. Μιλήσατε σε ό,τι αφορά για το ζήτημα της ασφάλειας των μεταφορών. Ένα σοβαρό ζήτημα. Αλήθεια. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ασφάλεια στις οδικές μεταφορές όταν από τη σχετική πρόταση για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των οδηγών εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι που μπορούν να δουλεύουν και 80 ώρες την ημέρα με αποτέλεσμα να αποτελούν δημόσιο κίνδυνο. Μιλάμε ότι στη φάση που διανύουμε, παρότι αυτή η Επιτροπή έκανε προσπάθειες, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, όχι με ευθύνη μας, αλλά από άλλους φορείς και από το Συμβούλιο αλλά και από τους πλειοκτήτες που πραγματικά δεν θέλουν να προσαρμοστούν ε, στα νέα, στο νέο καθεστώς, στα νέα στοιχεία ενισχυμένης ασφάλειας. Θέλω επιπρόσθετα με την ευκαιρία να πω ότι ένας άλλος στρατηγικός τομέας που έχει σοβαρή σημασία για εμάς είναι οι εσωτερικές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για τις οποίες η τελευταία έκθεση στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει συνταχθεί από την Επιστημονική Επιτροπή το 1999 δημοσιοποιήθηκε το 2002. Είμαστε δηλαδή 10 χρόνια χωρίς ένα εργαλείο το οποίο θα είναι πολύτιμο εφόδιο να ελέγξουμε πολιτικά πώς προχώρησαν αυτές οι πολιτικές αποφάσεις που πάρθηκαν σε ό,τι αφορά αυτούς τους τομείς. Παρότι κύριε Υπουργέ έχουμε, έχουμε κάνει επανειλημμένες ερωτήσεις τόσο προς την Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στους άλλους αρμόδιους φορείς μεταθέτουν τη δημοσιοποίηση της σχετικής έκθεσης από μήνα σε μήνα, από χρόνο σε χρόνο, από εβδομάδα σε εβδομάδα χωρίς μέχρι, μέχρι σήμερα να έχουμε ε, συγκεκριμένη απόφαση. Δεν θέλουμε να βγάζουμε αυθαίρετα συμπεράσματα. Θεωρούμε ότι τα στοιχεία που συγκροτούν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι πολύτιμο εφόδιο για τη δουλειά μας. Τέλος, θέλω να αναφερθώ ότι είναι σοβαρά τα προβλήματα που προκύπτουν και παραμένουν ανοιχτά σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Χρειάζεται αυτά τα ζητήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον να μπουν σε άμεση προτεραιότητα και να προευθυνθούν σε ό,τι αφορά τη συζήτηση γιατί ας μην γελιόμαστε μεταξύ μας βρισκόμαστε στην τελική φάση ολοκλήρωσης αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου και ό,τι προσπάθεια μπορεί να κάνει κάποιος σε αυτούς τους μήνες που έχουν αναπομείνει είναι ελάχιστη μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού του κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. il giro relativo ai... Τελείωσε ο πρώτος κύκλος των συντονιστών. Κύριε Υπουργέ, έχετε 10 λεπτά για να πρώτη σειρά απαντήσεων, μετά θα περάσουμε σε δεύτερο γύρο ερωτήσεων από τους συναδέλφους και μετά θα κλείσει πάλι ο Υπουργός. Eh, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μου υποβάλλατε. Ακούγοντας τις ερωτήσεις σας, θυμήθηκα όταν ήμουν και εγώ βουλευτής στην Τζεχία. Εδώ όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από τη χώρα μου, γιατί εκφράζονται πολύ διαφορετικές απόψεις. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, αλλά πρώτα απ' όλα θα σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας προς την ε, τσεχική προεδρία και την αυτοβιομηχανία που δεν είναι μόνο δικό μας. Δεν ξέρουμε ότι υπάρχει συνεργασία και εκ μέρους άλλων κρατών υποστηρίζουμε τέτοιο είδους συνεργασία και βεβαίως κανείς δεν θέλει να μετακομίσουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες και να γυρίσουν στη χώρα. Τόσο αφορά το πακέτο για τις αδικές μεταφορές, δύσκολα μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συνένεση η συνενετική λύση στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους για να καταλήξουμε σε λύση. Τόσο αφορά το καμποτάζ, πρέπει να πω ότι έχει γίνουν προσπάθειες και πάρα πολύ καιρό για να βρεθεί η λύση. Έχει επιτευχθεί πρόοδος, αλλά περιμένουμε και εσείς κάπως να μας βοηθήσετε. Ξέρω ότι η κυρία Τικάου και ο κύριος Γκρός έχουν έρθει ανεπιφήμως σε επαφή μαζί μας και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λογική συμβιβαστική λύση. Αυτό αφορά επίσης και τα ωράρια εργασίας. Ελπίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο, στο οποίο θα μπορέσουμε τελικά επίσης να καταλήξουμε συμφωνία. Όσον αφορά την Ευρωβινιέτ, το Ευρωπαϊκό Σήμα. Περιμένω τα αποτελέσματα των συζητήσεων σας. Ξέρω ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε κληρώσετε την έκθεση μετά την ψηφοφορία, μετά τις 60 και τόσο τροπολίες που Θα δούμε λοιπόν εμείς στο Συμβολίο ποια θα είναι η θέση στην οποία θα καταλήξετε. Είστε ε, σημαντικοί για το Συμβούλιο, όπως ξέρετε, και η άποψή σα είναι σημαντική. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα στα οποία εσείς θα καταλήξετε χωρίς να θέλουμε να προδικάσουμε τίποτε και να πούμε τίποτε εμείς αλλά προς το παρόν για το θέμα αυτό της Ευρωβινιέτ, το μπαλάκι είναι στο δικό σας το γήπεδο. Βεβαίω, και εμείς θα πρέπει να επομισθούμε τις ευθύνες μας για το θέμα αυτό και να καταλήξουμε σε κάποια λύση. Και βεβαίως τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Τώρα, όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα καταλήξει σε αποτελέσματα για το θέμα αυτό. Και πάλι η διαδικασία δεν είναι εύκολη, το θέμα δεν είναι εύκολο. Όπως ξέρετε είναι και από νομοθετικής πλευράς τα πράγματα πολύ στην Ευρωπαϊκή Θέληση, αλλά δεν θέλουμε να το παρακάμψουμε το θέμα. Θέλουμε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε λύση. Όσον αφορά τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, πιστεύω ότι οι θέσεις μας είναι συγκλίνουσες. Έχει επιτευχθεί μεγάλο μέρος της εργασίας εκ μέρους ημών και εκ μέρους της Επιτροπής. Και όντως φαντάζομαι ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες υπό τη δική μας Προεδρία να καταλήξουμε σε αποτελέσματα. Όλα εξαρτώνται από την πολιτική βούληση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Γνωρίζοντας όμως ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη θέση μας. Τώρα. Προσπαθώ να μην ξεχάσω κανέναν. Όσον αφορά την ερώτηση του κύριου Κράμερ. για θέματα αποζημιώσεων. Δεν ε, νομίζω ότι μπορώ τώρα να σας δώσω κάποια απάντηση. Αν θέλετε μπορώ να σας στείλω μία απάντηση γραπτός. Τώρα, το θέμα οδικές μεταφορές από τη μια σιδηροδρομικές από την άλλη. Το θέμα αυτό μπορεί να πάρει άπειρα χρόνια πριν διευθετηθεί. Εγώ σε επίπεδο περιφερειακής ε, διοίκησης, αν θέλετε, έπρεπε να ασχολούμαι όταν ήμουν στα πράγματα με το θέμα αυτό καθημερινά. Έπρεπε πάντα να έχουμε την ε, κατάλληλη νομοθεσία, τα κατάλληλα μέσα στη διαθεσή μας, <clears throat> διότι όλοι βεβαίως θέλουμε μέσω των μεταφορών να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες και κανένας δεν θέλει σε τέτοιου είδους θέματα να αποτύχει. Ως πολιτικός πιστεύω λοιπόν ότι ίσως ποτέ δεν θα λυθεί ικανοποιητικά για όλους το θέμα αυτό ειδικές μεταφορές από τη μια σύνδρομη για την άλλη. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε σοβαρά να βρούμε λύση. Τώρα, ίσως η κρίση που κάποιος μας κάνει να ενωθούμε. Μου αρέσει αυτή η τοποθέτηση διότι εδώ πρέπει κάτι να κάνουμε και να σταματήσουμε τα πολλά Όλοι στο ίδιο καράβι βρισκόμαστε τελικά. Και βεβαίως κανένας πλέον δεν έχει την πολυτέλεια να λέει ότι η οικονομική ανάψη χώρας του είναι 6 με 7%. Ξέρουμε ποια είναι και το πρόβλημα το οικονομικό των εθνικών κρατικών υπολογισμών και θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι με αποτελεσματικότητα. Σας ανέφερα προηγουμένω το Μάρκο Πόλο. Υπάρχουν και άλλα project που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα TNT, στον τομέα των μεταφορών και έχουν δοθεί αρκετά κονδύλια για να υποστηριχθούν τέτοιου είδους προγράμματα. Και βεβαίως γνωρίζουμε ότι αν προετοιμάσουμε καλά τα πράγματα και δοθεί, γίνει σωστά μία επένδυση, θα έχει και πάρα πολύ καλή αποδοτικότητα. Αυτό ελπίζω να το θυμάστε αύριο που θα ψηφίσει την Ευρωβινιέτ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω αυτή τη στιγμή εννέα γραμμένους στον κατάλογο για να μιλήσουν. Αν έχουμε δύο λεπτά ο καθένας, θα προλάβουμε. Πρώτος ο κύριος Μαρινέσκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας την προσοχή που αποδώσατε στις δύο εκθέσεις που το Κοινοβούλιο θεωρεί σημαντικές. Επίσης, σας ευχαριστώ για την πρόθεσή σας να οριστικοποιηθούν αυτές οι δύο εκθέσεις. Σας θυμίζω δόθηκε μία παράταση για την ψηφοφορία ακριβώς επειδή εσείς ζητήσατε περισσότερο χρόνο για να έχουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. ξεκίνησε ήδη μια σειρά συζητήσεων με τους κοιόδης εισηγητές και έχω να πω ότι εξής δύο τεινά. Καταρχήν, το πακέτο αυτό, οι δύο εκθέσεις μάλλον, θα εγκριθούν μαζί, ταυτόχρονα. Δεν θέλουμε να δοθεί αναβολή για το ένα από τα δύο, για μία από τις δύο εκθέσεις. Τώρα για ενδεχόμενε διαφορές που μπορεί να υπάρξουν μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά τον ενιαίο ουρανό, το Κοινοβούλιο θέλει να κλείνει το θέμα αυτό όσο πιο σύντομα γίνεται. Με συνθήκες μέγιστης ασφάλειας. Δυστυχώς όμως, μερικές τροπολογίες του Συμβουλίου δείχνουν την επιθυμία των κυβερνήσεων να παραμείνουν χωριστά όσο πιο πολύ γίνεται και να κρατήσουν τα πατροπαράδοτα τους προνόμια. Όσον αφορά για την υπηρεσία Οργανισμό για την Ασφάλεια, εμείς θέλουμε ο οργανισμός αυτός να πάρει ενεργότατο μέρος και στον έλεγχο του τι συμβαίνει μέσα στα κράτη-μέλη. Δυστυχώς όμως οι κυβερνήσεις θέλουν να πάρουν μια πιο μεγάλη φέτα από το γλυκό αυτό. Και η παράκλησή μου και των συναδέλφων υποθέτω παράκληση είναι να επιμείνετε στο συναδέλφο σας, να υποβάλλετε στο Συμβούλιο, να, μάλλον να, να παρουσιάσετε στο Συμβούλιο την κατάσταση ως έχει. Οι εκθέσεις έχουν στόχο την αύξηση της ασφάλειας της πτήσης. Δεν είναι μόνο για την αλλαγή του κλίματος Μιλάμε και για τα δικά μας ταξίδια, αυτά που κάνουμε, να γίνονται με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Άρα και οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν τον ίδιο στόχο, την ασφάλεια στις πτήσεις και, την, ε, και τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό του συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας άφησα να μιλήσετε λίγο παραπάνω επειδή είστε ένας από τους είσαι εισηγητές για το ένα στοιχεία του πακέτου. Παρακαλώ όμως άλλους συναδέλφους να μην ξεπερνάτε τα δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Μαρινέσκου, διότι είχαμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αντιλαμβάνουμε τι ελέγχθη, ότι όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν ένα πακέτο, πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα, είναι βασικά, αλλά αν ισχύσουν αυτό το οποίο υποθέτουμε σήμερα, δηλαδή ότι το Συμβούλιο θέλει να διαγράψει το ίμιση αυτού του πακέτου, και να διαγράψει το ίμιση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε δεν θα συμβεί τίποτα και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρξει πλειοψηφία σε αυτό το κοινοβούλιο για να στηρίξει μια τέτοια λύση ε, διότι ε, πρέπει να συζητήσουμε τις ε, αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Αεροπλοείας και αντιλαμβάνομαι γιατί ορισμένα κράτη δεν θέλουν ε, να χρειαστεί να ελέγχεται η ε, αρχή τους ε, της αεροπλοείας αλλά για την Ευρώπη κάτι τέτοιο επιβάλλεται και θα πρέπει να καταλήξουμε σε μία λογική συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σήμα θα είχα την τάση εδώ να ξεκινήσω μία συζήτηση και να σας πω ότι ε, ο θόρυβος και ε, οι εκπομπές ε, όπως τις παρουσιάζει ο κύριος Γιαρζεμπόφσκι δεν κάθομαι τυχαία στην άλλη άκρη της σειράς από τον κύριο Γιαρζεμπόφσκι αλλά το ερώτημα είναι ποιες είναι εδώ οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ κρατών μελών ποια είναι τα κράτη που το επιθυμούν λίγο ποιοι είναι αυτοί που το θέλουν πολύ και ούτω καθεξής. Και το τρίτο ερώτημα, σας, ε, δεν απαντήσατε στην ερώτηση του κυρίου Κράμερ σχετικά με τα τεράστια επιβατικά, διότι ξέρω ότι υπήρξε μία συζήτηση και κάπου θα έπρεπε να υπάρχει και μία δέσμευση. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε γνώμη κάθε χρόνο. Γιατί ε, ε, ε, πιστεύετε ότι θα προχωρήσει αυτό το θέμα και ποια είναι η θέση του Συμβουλίου επ' αυτού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Μεταφορών Μπέντλ, είπατε ότι έρχεστε από μία από τις δέκα περιοχές της Ευρώπης που έχουν τις περισσότερες μεταφορές, αλλά και εκεί χρειάζεται να μειωθεί η κίνηση. Εάν λοιπόν πάρουμε στα σοβαρά την στρατηγική της Λισαβόνας, όπου η ανάπτυξη των μεταφορών πρέπει να διαχωριστεί από την οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να δούμε πού μπορούμε να μειώσουμε τις μεταφορές, πού υπάρχουν μεταφορές που δεν αποδίδουν σε ε, κανένα προσόν. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Επίσης σχετικά με τα ερωτήματα που θίξατε για την ασφάλεια των μεταφορών ε, έχουμε μία συγκεκριμένη απέτηση για τη Βόρεια Ιταλία για ένα κομμάτι του, ε, του, του αυτοκινητοδρόμου που δεν επιτρέπεται να περνούν τα φορτηγά το ένα το άλλο διότι ε, έτσι θα μειώσει κανείς κατά 30% ε, τα δυστυχήματα που προκαλούν αυτές οι υπερβάσεις. Αν λοιπόν ε, θέλουμε να μεταβιβάσουμε τις μεταφορές από το αυτοκίνητο στο σιδηρόδρομο θα πρέπει να ε, αποσύρουμε τα παλιά, ε, τους παλιούς σειρμούς για να μπορέσει κανείς να έχει σύγχρονο εξοπλισμό. Διότι από τη Γερμανία ναι μεν έχουμε σύγχρονα οχήματα αλλά από την Ιταλία έχουμε πολύ παλιούς σειρμούς και ακόμα ακόμη, ε, και ακόμη και αυτοί οι οποίοι είναι κατά των σιδηροδρόμων αναγκάζονται να τα χρησιμοποιούν. Επίσης ο κύριος Ταγιάννη ε, μας είχε πει ότι το θέμα τώρα είναι στο Συμβούλιο. Δηλαδή μετά από 10 χρόνια θα μπορέσει τέλος πάντων να ολοκληρωθεί αυτή η διεργασία και να περάσει αυτή η νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σήμα Κυκλοφορία. Δεν είναι ε, το θέμα ότι ο κύριος Γιάννης έχει προσωπικά ένα πρόβλημα. Δεν συμβαίνει αυτό. Το κόστος για την εισαγωγή του ευρωσήματος είναι μεγάλο. Είναι δεδομένο και μεγάλο. Τα ωφέλη όμως για την μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα είναι συζητήσιμα. Και ρωτώ, κύριε Υπουργέ. Η Κομισιόν πρόσφατα παρουσίασε ένα σχέδιο κανονισμού για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα μεταφορών φορτίου με τους σιδηροδρόμους. Υπάρχουν όμως μερικά προβλήματα σε σχέση με αυτή την πρόταση. Γι' αυτό μερικά κράτη λένε όχι στην πρόταση αυτή μέχρι στιγμής. Εσείς, ερωτώ, σκοπεύετε να πάρετε μια πολιτική πρωτοβουλία για να βρεθεί συμβιβασμό. Πρόεδρος. Παραμένει η ερώτηση λοιπόν προς τον κύριο Υπουργό. Συνεχίζουμε τον συνάδελφο Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον κύριε Προεδρεύοντα διότι βρισκόμαστε στο τέλος της θητείας μας. Και εσείς, στο τέλος του Ιουνίου, ολοκληρώνω την Προεδρία σας. Η κρίση όμως δεν θα τελειώσει. Τι θα κάνετε λοιπόν για να κάνετε κάτι και στις οδικές μεταφορές και στα όλα τα παλιά οχήματα που κυκλοφορούν. Επίσης, τι θα κάνετε για να μπορέσετε να βελτιώσετε και την ασφάλεια σε όλους τους ε, τομείς ε, των μεταφορών και στις αεροπορικές και στις και στις οδικές μεταφορές. Τι θα κάνετε για την ασφάλεια των πολιτών. Δεν θα υπάρχει κοινοβούλιο σε λίγους μήνες, κάτι πρέπει να κάνετε όμως, διότι εσείς θα μείνετε μόνοι σας. Τώρα, επίσης, <clears throat> τι προβλέπετε να γίνεται με τον διάδρομο ο οποίος θα ενώσει την Σουηδία, την Πολωνία, την Τσεχία με την Νότια Ευρώπη. Θέλετε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, σας ευχαριστώ που είπατε ότι οι δαπάνες για να βελτιωθούν οι υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Κυρίως σε εποχή κρίσης. Ε, εμείς όμως θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί περιορίζοντας τις δαπάνες στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Φούλα. Κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα και εγώ να θέσω το θέμα της οδικής ασφάλειας. Όντως, βρισκόμαστε στο 2009 και ο στόχος που τέθηκε το 2010 ήταν να μειωθούν κατά το 50% οι θάνατοι στους δρόμους της Ευρώπης. Πώς νομίζετε ότι μπορείτε να υλοποιήσετε το στόχο αυτό ή να τον προσεγγίσετε στο μέτρο του δυνατού. Και πιο συγκεκριμένα, ποια είναι η στρατηγική σα για να καταλήξετε σε συμφωνία για το κείμενο το οποίο ψηφίστηκε στι 17 Δεκεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ενισχυθεί σε θέματα οδική ασφαλεία η διασυνοριακή συνεργασία. Δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα για το κείμενο αυτό σε επίπεδο ε, Σύμβουλου Υπουργών. Θα ήθελα λοιπόν γι' αυτό κυρίω το θέμα να επιστήσω την προσοχή σα και να ζητήσω απάντηση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη γιατί άρχισε το αεροπλάνο μου, έφτασα αργά και να πω στον κύριο Πρόεδρε ότι δεν έχουμε μόνο αντιπαραθέσεις και μονολυθικές ακραίες θέσεις ο καθένας μας. Όπως ξέρετε η Ευρώπη είναι κάτι το πολύ πολύπλοκο. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα λυθεί το πρόβλημα. Ξέρετε όμως ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα με την πρόταση που έκανε η Κομισιόν. <clears throat> Τώρα για θέματα συμφόρησης. Κύριε Υπουργέ, η λύση προς την οποία εμείς οδηγούμεθα μπορείτε να μας βεβαιώσετε από τις συζητήσεις που είχατε στο Συμβούλιο ότι δεν έχει ασάφειες. Τώρα, την Ισπανίθια από το εξή. Ξέρω ότι στο Συμβούλιο υπάρχει πρόβλημα, πρόβλημα σε σχέση με τις διάφορες ρήτες τις οποίες μπορέσαμε εμείς να προωθήσουμε για θέματα ασφάλειας των αεροπορικών των αερομεταφορών, αλλά δεν ξέρω τι συνέβη, κυρίως με τον ε, γραμματέα του συμβολίου. Δεν ξέρω τι ακριβώ συνέβη, αλλά εν πάση περιπτώσει τα θέματα της ασφάλειας των αερομεταφορών, κυρίως στο Γιβλαρτάρ, είναι θέματα με τα οποία εμείς έχουμε ασχοληθεί πολύ και προσφέρουμε λύσεις. Βασιστείτε λοιπόν στο δικό μας κείμενο και όχι σε αυτό του συμβουλίο για το οποίο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, σε σχέση με τις ε, ασφάλειες γενικά των ειδικών μεταφορών. Όπως είπε η κυρία Φουρέ, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Σε πρώτη ανάγνωση του σφαιρικού προγράμματος της ε, τσεχικής προεδρίας απογοητεύτηκα γιατί εδώ το μόνο που εμφανιζόταν ήταν πρόταση για νέο πρόγραμμα ασφάλειας των οδικών μεταφορών από το 2011 και μετά. Πριν να προχωρήσουμε όμως εκεί θα πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα Πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον στόχο τον οποίο θέλουμε να υλοποιήσουμε μέχρι το 2010, δηλαδή να μειωθεί στο 50% ο αριθμός των ε, θανάτων από αυτοκινητικά ατυχήματα. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι κάνετε εσείς για αυτό το θέμα. Εμείς σας δώσαμε μία σαφή κοινοτική λύση πρώτου πυλώνα, αλλά μέχρι τώρα οι λύσεις που προβλέπονται από το Συμβούλιο αφορούν τον τρίτο πυλώνα. Ξέρουμε ότι σε περίπτωση διμερών συμφωνιών οι συμφωνίες πλαίσιο δεν προσφέρουν λύση και θα θέλαμε να προχωρήσετε σε κάποια πιο αποτελεσματική λύση, κυρίως εάν εγκριθεί και η νέα συνθήκη. Σας παρακαλούμε λοιπόν, επειδή είστε νέος, εσείς όπως λέτε, αφήστε πίσω τα προβλήματα του παρελθόντος και με μεγάλο θάρρος προσπαθήστε να προσεγγίσετε τη θέση του Κοινοβουλίου που είναι και η θέση της πλειοψηφίας των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Προεδρία για την συνεργασία και για την ε, πρόθεση συμβιβασμού στις τριμερείς διαλόγους, πράγμα το οποίο θα χρειαστεί να ε, διέπει και τη συζητήσεις των επομένων εβδομάδων για τις οδικές μεταφορές. Έχω να πω τα εξή για τις οδικές μεταφορές. Ο κανόνας των 12 ημερών μας ενδιαφέρει όπως είπαν συνάδελφοι. Επίσης πιστεύουμε ότι ε, δεν ε, αναφερόμαστε εδώ μόνο εις ε, τις συνήθειες στα διάφορα κράτη αλλά ότι η ασφάλεια έχει σημασία για τις 12 ημέρες και επίσης θέλω να υπάρχει συνέπεια για το καμποτάζ περιορίστε την αγορά και με εκπλήσει γιατί υπάρχουν αντεφατικές δηλώσεις και διαπίστωσα ότι το Ενωμένο Βασίλειο ζητά ε, ένα περιορισμό της αγοράς και καλύτερη ρύθμιση, δηλαδή ολόκληρες χώρες αλλάζουν γνώμη και πέραν αυτού εσείς εδώ ζητάτε ένα περιορισμό γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνετε κατόπιν ετήσεως του Συμβουλίου ακόμη και αν δεν συμφωνείτε. Αλλά ε, κατά τη γνώμη μου έπρεπε να είναι κανείς ανοιχτό προς το μέλλον. Δηλαδή δεν μπορούμε σήμερα να περιορίζουμε την αγορά και να μην ε, συνδυάζουμε το άνοιγμα με ορισμένα κριτήρια και για να υπάρχει συνέπεια Πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατόπιν προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε αναφερθεί εις ε, τις ε, σκιώδεις εγκαταστάσεις, δηλαδή στις εταιρείε μαϊμού, δηλαδή αυτές οι οποίες ναι. βρίσκονται σε χώρες, οι οποίες για κοινωνικούς ε, ή φορολογικούς λόγους προσφέρουν προσόντα που στρεβλώνουν την αγορά. Αν δηλαδή κανείς προσπαθεί να βελτιώσει την ασφάλεια και επιτρέπει αυτές τις σκιώδεις έδρες, τότε ε, δεν θέλω να μου απαντήσετε από αυτού σήμερα, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι για τη δικιά μας άποψη το θέμα αυτό είναι στενά συνδεδεμένο με το μέλλον του τομέα. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι θέλουμε προσωρινά να προστατεύσουμε την αγορά και από την άλλη, ε, φορά, από την άλλη πλευρά με έδρες στο Λουξεμβούργο που είναι μια πολύ συμπαθητική χώρα. Ε, θα ήθελα να ήξερα πόσα φορτηγά αυτοκίνητα χωράνε σε ε, μια ταχυδρομική θηρίδα που είναι όλη η έδρα αυτής της εταιρείας. Λοιπόν, ε, εάν ε, υπάρξουν τέτοιοι περιορισμοί πρέπει να δούμε αν είναι συνεκτικοί και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι πάντοτε έχουμε πρεσβεύσει την επικουρικότητα σύμφωνα με τις αρχές της ασφάλειας και της υποδομής για κάθε χρόνια, κάθε, για κάθε χώρα η οποία θα έπρεπε να μπορεί να αποφασίζει αυτό τελώς. Ελπίζω ότι δεν έχω ε, ξεχάσει κάποιο θέμα, αλλά πιστεύω ότι αυτά είναι η άποψη της πλειοψηφίας. Δηλαδή ε, το Κοινοβούλιο δεν ήθελε να ρυθμίσει τα πάντα, άφησε πολλά στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ε, κλείνει ο κατάλογος με τον κύριο Στόκμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Θέλω να θίξω και δύο άλλα θέματα τα οποία αναφέρατε. Είπατε ότι κατά την κρίση θα έπρεπε να συσπηρωθούμε πολιτικά και δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό και επίσης η κρίση έχει θέματα στην ε, νομοθεσία μας ε, τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί και θέλω να σας υπενθυμίσω. Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα Μαρκοπόλο διότι εκεί ε, θέλουμε να προχωρήσουμε για να υπάρξει μια πιο γρήγορη διεκπαιρέωση και να συμφωνήσουμε με τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρόλο που πιστεύω ότι αν αυξήσουμε τις ε, ε, παροχές, ε, μειώσουμε τα δικαιώματα και δημιουργήσουμε νέα γραφεία, επιβαρύνουμε πολύ το σύστημα. Αλλά καλό θα ήταν να έχουμε καταρχήν μία ανάλυση και θα ήθελα να σχολιάσω το εξής. Στην περίοδο της κρίσης έχουμε μία μείωση και μεταφορά των μεταφορών προς τις οδικές μεταφορές και ορισμένα από τα προγράμματα τα οποία εδώ προσπαθούν να μετακτοπίσουν τον τρόπο μεταφοράς δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν και θα διακινδυνεύσουν. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε αν σε περίοδο κρίσεως την οποία θα πρέπει να οριοθετήσουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτά τα προγράμματα χωρίς να τα καταστρέψουμε, διότι πρέπει να μεταφερθούν οι μεταφορές από το ένα μέσο στο άλλο. Επίσης σχετικά με τις ρυθμίσεις και την ομοθεσία, όπως έγινε για την 10 η Σεπτεμβρίου, δεν θα έπρεπε να ξέρει κανείς πώς κατανείμει τα σλότ, πώς ε, τα οργανώνεις, διότι θα ήταν κακό εάν αεροπλάνα τώρα στην, ε, ε, στην κρίση εξυπηρετούν τα σλότς και διακινούνται με άδεια αεροπλάνα απλώς για να κρατήσουν τα σλότς, τις θέσεις δηλαδή που έχουν γιατί αυτά έχουν κάποιο φορολογικό προσόν. Δηλαδή θέλουμε να κατευθύνουμε την ε, βιομηχανία αυτή σε τόσο λαθασμένη κατάσταση, ε, κατεύθυνση σε περίοδο κρίσεως. Και βλέπω ότι υπάρχουν ε, δύο θέματα τα οποία πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε πώς η κρίση επηρεάζει τα προγράμματά μας και κατά τα άλλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και έχετε όντως καταρτήσει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωράει χωρίς να λάβουν υπόψη ότι έχουμε εκλογές. Τώρα προσπαθούν να περάσουν θέματα αποζημιώσεων πολύ γρήγορα και θα ήθελα να σας πω ότι δεν συμφωνούμε με αυτό το σύστημα αλλά αυτό θίγει και εσάς. Σας φορτώνουν με τόσα πράγματα, ώστε δεν μπορείτε πλέον ούτε να προετοιμαστείτε σωστά, ούτε να διεκπαιρώσετε όλα τα θέματα. Θα ήθελα όμως να μου πείτε αν στα δύο αυτά σημεία δεν θα έπρεπε ίσως να αλλάξουμε κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε με το δεύτερο γύρο και τελευταίο και θα δώσουμε την ευκαιρία στον προεδρεύοντα να σχολιάσει ένα σωρό διαφορετικά θέματα. Βέβαια υπάρχει μια αντίφαση εδώ εσωτερική δική μας. Του ζητάμε, του ζητήσαμε μάλλον στην αρχή να, την ε, συγκεντρώσει την προσοχή σε ορισμένα σημεία και μετά υποβάλαμε ένα σωρό διαφορετικές ερωτήσεις και δεν είναι δυνατόν να δώσει απάντηση σε όλες. Είμαι σίγουρος ότι θα βάλει τα δυνατά του και του δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσο πιο πολλές ερωτήσεις μπορέσω. Αν δεν ε, είμαι σε θέση να απαντήσω σήμερα, θα σας δώσω την απάντηση αργότερα. Παίρνω τις ερωτήσεις με τη σειρά. Μερικέ φορέ μπορεί να έχω πρόβλημα με το πώ προφέρω τα ονόματα. Ζητάω προ, προκαταβολικά συγγνώμη. Αρχίζω με τον κύριο Μαρινέσκου. Αναφερθήκατε στην ανάγκη να συζητηθεί ο ενιαίος ε, Ευρωπαϊκός Ουρανός και η ΆΣΑ. Έπρεπε και τα δύο θέματα αυτά να συζητηθούν ταυτόχρονα. Και θα συμβεί αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε το χρόνο που χρειαζόμαστε, όπως τον ζητήσαμε προκειμένου να συζητήσουμε μερικά εσωτερικά θέματα που εμείς είχαμε και είχαμε τώρα το χρόνο σιγά σιγά να τα χωνέψουμε. Είναι πολύ δύσκολο να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο σημεία. Πρέπει να τα πάρουμε ταυτόχρονα. Και πιστεύω ότι τώρα υπάρχει κοινή θέση στο Συμβούλιο. Η ερώτηση του κυρίου Λάικφριντ, αν προφέρω σωστά το όνομα, ζητάω και πάλι συγγνώμη, για τα φορτηγά. Εν μέρη απαντήσατε ο ίδιος στην ερώτησή σας. Είναι τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για αυτού του είδους τα, τα οχήματα. Ίσως να υπάρξει κάποια μέρα μια απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Ευρωκοινοβούλιο, τότε θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια λύση για τα trailers, για τα trailers. Προς το παρόν όμως είναι ένα θέμα πάρα πολύ ε, λεπτό όσον αφορά τις κυβερνήσεις ευρωσήμα, ευρωβινιέτ. Τι διαφορές υπάρχουν. Ήδη αναφέρθηκε, το είδαμε στη συζήτηση, η πιο μεγάλη διαφορά είναι η στάση των χωρών διαμετακομιστικού εμπορίου σε σχέση με χώρες που δεν θεωρούν τον εαυτό τους διαμετακομιστικές χώρες ή που βρίσκονται στην περιφέρεια. Να βρεθεί μια κοινή γλώσσα ανάμεσα σε αυτά τα δύο στρατόπεδα, αυτό είναι το πιο μεγάλο ζητούμενο όσον αφορά το ευρωσήμα. η σιδηροδρομική διάδρομη. Ο κύριος Κούστασερ με ρώτησε. Απαντώ. Συμφωνούμε ότι οι διάδρομοι έχουν προτεραιότητα και για μας. Έχει ιδιαίτερη ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την κινητικότητα των ανθρώπων και όσον αφορά τις διάφορες κρίσεις που ζούμε. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Όχι μόνο μεταξύ βορρά-νότου και ανατολής-δύσης, Πραγματικά και οι δύο αξονες είναι σημαντικοί. Βορρά νοτος Ανατολή Δύση. Και οι δύο είναι σημαντικοί. Το είπα και στην εισαγωγή μου. Ο κύριο Ντιχόνη ρώτησε για την ανταγωνιστικότητα μεταξύ δρόμων σιδηροδρόμων. Συμφωνούμε, ξέρουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι σε σχέση με την οδική μεταφορά επιβατών και με τη μεταφορά με το τρένο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το πώς θα βελτιώσουμε τη μεταφορά των επιβατών. Κύριος Λιμπεράτσχη, διάδρομοι DNT. Και τα διόδια τα οποία πληρώνονται, οι διάφορα τέλη. Δεν είμαι κάπως ασαφής στις σημειώσεις μου. Κάποιος, κυρίως και κυρία βουλευτές ρώτησαν για την οδική ασφάλεια και οι δυο τους αναφερθήκατε, δυο σας, αναφερθήκατε στο θέμα του κανονισμού για την ασφάλεια όσον αφορά διασυνοριακά θέματα. Όσον αφορά την αρμοδιότητα υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη μεταξύ των μεταφορών από τη μια μεριά και των εσωτερικών θεμάτων και θεμάτων δικαιοσύνης από την άλλη. Μιλάει για δύο διαφορετικά υπουργεία δηλαδή. Πρώτα θα πρέπει να δούμε πού υπάρχει επικάλυψη στις αρμοδιότητες. Αν δεν το κάνουμε αυτό προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε. Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα ποιο Υπουργείο είναι κυρίως το υπεύθυνο. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί μια για πάντα. Γιατί όπως αυξάνεται και διευρύνεται το δικό δίκτυο, έχουμε όλο και περισσότερες ε, διασυνοριακές κινήσεις και προβλήματα. Αυτά για το θέμα της ασφάλειας. Αυτό θα συζητηθεί στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών του Απριλίου. Ο κύριος Γκρός αναφέρθηκε στον κανόνα των 12 ώρων. Νομίζω ότι σωστά το πιάσατε το θέμα. Και εμείς θέλουμε να πετύχουμε ένα συμβιβασμό. Μία δυνατότητα βρίσκεται στο καμποτάζ σε σχέση με τον κανόνα των 12 ωρών. Μπορεί να πετύχουμε κάτι προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν συμφωνήσουμε ή όχι. Οι διάφορες ε, πλασματικές εταιρείες Αυτό είναι θέμα της αγοράς πώς κινείται η αγορά. Θα το συζητήσουμε στο Συμβούλιο. Θέλουμε να αποφύγουμε ορισμένα πράγματα ως νομοθέτες. Εγώ δεν εκφράζω εδώ τις απόψεις της Τσεχίας, αλλά του Συμβουλίου συνολικά. τις απόψεις της πλειοψηφίας του Συμβούλιο, πιο συγκεκριμένα. Άσχετα ποια είναι η προσωπική γνώμη του Τσέχου Υπουργού. Διότι παίζεται το κύρος της τσεχικής προεδρίας στο σημείο αυτό. Μάρκο Πόλο. Ο κύριος Στόκμαν. Είπατε ότι τα μεταφερόμενα προϊόντα σε ποσότητα μειώνονται. Υπάρχουν, υπήρξαν πολλά, πολλά υποσχόμενα οικονομικά προγράμματα όταν ξεκίνησαν, γιατί ο προγραμματισμό είναι συνήθω πολιετή. Ποτέ δεν προβλεπότανε ότι θα έχουν αυτά τα σοβαρά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης που ζούμε. Αυτό πρέπει και η Ένωση και τα κράτη-μέλη να το αντιμετωπίσουμε δεν είναι όμως κάτι που αφορά αποκλειστικά τις μεταφορές. Αφορά οποιοδήποτε κλάδο όπου έχουν γίνει επενδύσεις. Ευχαριστώ που αναφερθήκατε στο θέμα του να δοθούν σλότ σε αεροπορικές εταιρείες. θα το χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που είπατε στη συζητήση στο Συμβούλιο. Δεν είμαι καταρχήν αντίθετος. Και με αυτό ελπίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις. Αν όμως, και είναι πολύ πιθανό, αν όμως υπάρχουν ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν, να θα σας δώσω εξηγήσεις είτε γραπτός, είτε διμερός, είτε εδώ, είτε στην Τσεχία. Είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και για την ευγενή σας στάση. Μη πάρα και Πρόεδρος. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τις σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί μεταξύ Τσεχικής Προεδρίας και της Επιτροπής μας. Έχουμε μια αντίφαση. Θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και ταυτόχρονα ε, δεν έχουμε χρόνο για να καλυφθούν όλα τα θέματα τα οποία αναφέρουμε. Το ίδιο θα συμβεί και σε αυτό το εξάμεινο. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι θα σημειωθεί και πρόοδος και διαβεβαιώνω ε, εκ μέρους όλων των συναδέλφων τον Προεδρεύοντα ότι το Κοινοβούλιο θα έχει την ίδια υψηλού επίπεδου συμπεριφορά απέναντί σας όπως είχαμε και στο παρελθόν. Προκειμένου να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από κοινού για τα δύο θεσμικά όργανα που πουμε δυο Δύο-τρία λεπτά να συνοδεύσω τον Υπουργό έξω και συνεχίζουμε.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 Please may the meeting come to order. We continue our uh, meeting. Uh, We want to ex- talk and discuss. Συνεχίζεται η Έχουν τους όπως με τους αρμόδιους για τη ΣΤΟΑ, κυρία Μπάρση Πατάκη. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι είναι σύντομοι. Πείτε μας καταρχήν τις απόψεις πώς έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής. Η κυρία Μπάρση Πατάκη πρώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω σήμερα να αναφερθώ σε δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στα πλαίσια της Επιτροπής ΣΤΟΑ. Καταρχήν είναι το θέμα της ναυσιπλοείας και δεύτερον ε, το θέμα των οδικών μεταφορών. Καταρχήν όσον αφορά τα δίκτυα ε, έγινε ένα συνέδριο την 1η ε, Σεπτεμβρίου του 2006 και ένα εργαστήριο το οποίο οργανώθηκε εν ονόματι της ε, Επιτροπής ΣΤΟΑ οργανώθηκε από τον καθηγητή Γκιούντερ Χάιμ από το Μόναχο με πολύ ψηλά ιστάμενους εμπειρογνώμονες που παρουσίασαν τις απόψεις τους σχετικά με το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Ε, εκεί υπήρχε μία σαφής δήλωση για τη σημασία του προγράμματος και τη σημασία των εφαρμογών. Ελέγχθη ότι το πρόγραμμα Αγκαλιλαίο μπορεί να ευθυγραμμιστεί με την ανάπτυξη των κινητών τηλεφώνων. Θεωρείται ότι 150.000 θέσεις μπορούν να δημιουργηθούν μέσω του προγράμματος Γαλιλαίο και οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι το ποσοστό αυτό θα, ε, ε, θα αυξηθεί με την δημιουργία θέσεων στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες. Ε, για το 2025 η ομάδα προβλέπεται ότι θα έχει ένα προϋπολογισμό εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Επειδή λοιπόν αυτό το εργαστήριο οργανώθηκε πριν από δύο χρόνια, υπάρχουν ορισμένες πολύ σημαντικές απόψεις οι οποίες καλό θα ήταν να τονιστούν και σήμερα. Δηλαδή, εκείνη την εποχή όλοι ξέραμε ότι τον Καλλιλέο καθυστερούσε και το σύνολο του αστερισμού σχετικά με τους δορυφόρους επρόκειτο να καθυστερήσει και να ολοκληρωθεί γύρω στο 2010. Τώρα ξέρουμε ότι ενδέχεται αυτό να καθυστερήσει ως το 2013. Συζητήθηκε λοιπόν κατά τη διάρκεια του workshop ποια θα ήταν η διαδικασία για την ανάθεση των, των σταθμών αυτών και τα πρότυπα τα οποία έπρεπε να επεξεργαστούμε. Το βασικό, η βασική αρχή ήταν η κατανομή των κινδύνων και ήταν προφανές ότι ορισμένοι από τους κινδύνους θα αναλαμβάνονταν από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή ε, οι ε, υπερβάσεις κόστους, η ολοκλήρωση, αλλά ε, υπήρχαν πολλά ερωτήματα σχετικά με την αστική ευθύνη, με την, ε, ε, τις καθυστερήσεις και τις υπερβάσεις του κοστολογίου και γι' αυτό χρειάστηκε να αλλάξει το πρότυπο χρηματοδότησης του Γαλιλαίου το χρονοδιάγραμμα είναι πιεσμένο. Δεν αναφέρεται μόνο στην ανάπτυξη του προγράμματος Γαλιλαίο, αλλά αναφέρεται επίσης και στο ρυθμιστικό περιβάλλον, διότι υπάρχουν πολλοί φόβοι για τις εφαρμογές και για διάφορα άλλα θέματα τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμη όπως παραδείγματο χάρη οι ρυθμισμένες υπηρεσίες που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος. Υπάρχουν ευαίσθητα θέματα όπως η προστασία των δεδομένων και η, ε, η κάλυψη της ε, ιδιωτικής ε, ε, ταυτότητος τα οποία έπρεπε να ληφθούν υπόψη και υπήρχαν και άλλα θέματα που έπρεπε να σκεφτούμε. Για να υπάρχει ε, μία μικρή μεταβατική περίοδος από τη μία φάση στην άλλη έπρεπε να γίνει κατανομή των ευθυνών και, της, και κατανομή ε, των κινδύνων μεταξύ ε, του ιδιωτικού και δημοσίου τομέως και το πρόβλημα αυτό υπάρχει και σήμερα και με το τέλας. Ε, το ίδιο, τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν δηλαδή και σήμερα και δεν έχουν επιληθεί ακόμη. Άρα το σεμινάριο αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον διότι τόνισε ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε το Γαλιλαίο. Η δεύτερη λύση ήταν η εναλλακτική λύση για οδικίες και αεροπορικές μεταφορές και ο εισηγητής ήταν ο Μάρκο Χάμπορν. Μία ευρεία επιλογή ε, έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες και ορισμένες τεχνολογίες ήδη έχουν τεθεί στο εμπόριο. Αλλά δεν είναι δυνατόν να σκεφτούμε ποιες θα είναι οι τεχνολογίες οι οποίες θα υπερισχύσουν στην Ευρώπη και άρα προσπαθούμε να καταρτήσουμε έναν κατάλογο με ε, προσφορές και μία επισκόπηση των ε, εναλλακτικών λύσεων που υπάρχουν για τις οδικές και τις αεροπορικές μεταφορές. Το δε συμπέρασμα ε, αυτής της μελέτης είναι ότι όλοι οι εμπειρογνώμονες συμφώνησαν ότι είναι υπεύθυνοι για τις συζητήσεις για εναλλακτικά καύσιμα, αλλά υπάρχουν τρία βασικά θέματα. Καταρχήν, η πνόγνωση για μείωση ε, ή εξαφάνιση των ε, ορυκτών καυσίμων, ε, τα ανταγωνιστικά ωφέλη, η ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων και το βασικό, το βασικό συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι έχουμε καλές πιθανότητες να λύσουμε το πρόβλημα σχετικά με τον οδικό τομέα, αλλά έχουμε σοβαρά προβλήματα ε, όσον αφορά τον αεροπορικό τομέα. Και η κατάσταση είναι τέτοια, ώστε στις αεροπορικές μεταφορές υπάρχει πολύ αυστηρή ρύθμιση σχετικά με την ασφάλεια και δεν είναι εύκολο να βρεθεί μία σωστή λύση. Οι τεχνολογίες οι οποίες συγκεντρώνονται στο κατάλογο είναι πολύ, πολύ καλές αλλά όλες παρουσιάζουν και προβλήματα και κάθε τεχνολογία αντιμετωπίζει σχολίες όσον αφορά την κάλυψη της μελλοντικής ζητήσεως από Ευρώπη των 27. Συνάδελφοι, έχω πάρα πολλά να σας πω για το, ακόμη για αυτό το ε, εργαστήριο και αν θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ κυρία συνάδελφε και τώρα δίνω το λόγο εις ε, τον επόμενο μιλητή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. έχοντας ακούσει τη συνάδελφος και συνεχίζοντας θα πω το εξής υπάρχουν δύο θέσει αλλά ήδη υπάρχουν και δύο άλλε εκθέσει για το θέμα αυτό, τις οποίες έχουμε ξεχαστεί εδώ και καιρό. Πρώτα απ' όλα, στον τομέα των μεταφορών, πρώτα απ' όλα έχουμε το θέμα της ασφάλειας στα τούνελ και δεύτερον, ένα δεύτερο θέμα που αφορά το μέλλον των μεταφορών ε, ε, μικρής διάρκειας στην Ευρώπη. Λοιπόν, ασχοληθούμε με το πρώτο. Η ασφάλεια στα τούνελ. Πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά βιβλικό και τεχνικό. Μπορέσαμε να αναλύσουμε διάφορα συμβάντα και ατυχήματα στα διάφορα τούνελ στις σύραγγες της Ευρώπης από το 1995. με ανάλυση των κινδύνων σε όλες τις ε, φάσεις της σύλληψη, ε, της ε, δημιουργίας αυτών των σεργών και ο στόχος μας είναι να κάνουμε κάποιες συστάσεις ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης κάποιων από τα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν σε περίπτωση ατυχημάτων, δυστυχημάτων, βασιζόμενοι κυρίως στα πορίσματα στα οποία κατέληξαν οι εμπειρογνώμων. Δεν υπάρχει βεβαίως κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά στη μελέτη που έγινε βλέπουμε ποιες είναι οι διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την ανάλυση των κινδύνων στις ευρωπαϊκές σύραγγες. Γίνεται λόγος για τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε για να κάνουμε την ανάλυση του κινδύνου και πώς τα αντιμετωπίζουμε σε όλα τα επίπεδα. Πρόληψη τη στιγμή της ε, σύλληψης της ιδέας κατασκευής μιας τέτοιας σύνδεξης. Βεβαίως, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, ιδιαιτερότητες και το γεγονό ότι εξελίσσονται τα πράγματα και σε θέμα ακόμη και για τις σύραγγες. Και Βεβαίω με τα τρένα μεγάλη ταχύτητα, επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρέπει να γίνουν διάφορες αναπροσαρμογές και στη συναγγίση. Θα πρέπει στο μέλλον λοιπόν να γίνει μία ανάλυση κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υπάρχει προσέγγιση κοινή για όλους. Δεύτερο θέμα, και εδώ πάλι θα πω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, δεύτερος φάκελο. η μεταφορές με προοπτική στην Ευρώπη μακροπρόθεσμη, δηλαδή το 2050. Πρέπει να πω ότι έγιναν συζητήσεις πολύ ενδιαφέρουσες την ε, παρουσία εμπειρογνωμόνων σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση, σε δεύτερο στάδιο. Θελήσαμε να μελετήσουμε κατά κάποιο τρόπο τη θέσπιση ενός εφόρου συστήματος το 2050 με, την, ε, τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων. Δηλαδή, να εξαρτώμεθα λιγότερο από την ε, κατανάλωση καυσίμων, να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Βεβαίως οι στόχοι μας ήταν πολύ μεγάλη επίβολη, είχαμε μιλήσει για μειώσει από το 60%, ενώ ξέρουμε ότι συγχρόνως δεν θα πρέπει να μειωθούν τα ποσοστά πρόσβασης σε αυτό το είδος μεταφορών. Προβλέπονται τρεις δυνατότητες εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προσπαθούμε συγχρόνως να απαριθμίσουμε τα πέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους τους οποίους θέσαμε. Τρεις δυνατότητες. Μία ισχυρή και πολύ καλά οργανωμένη Ευρώπη. που θα κάνει σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των τεχνολογιών εχμής για να είναι αποτελεσματική. Δεύτερο σενάριο, μια Ευρώπη λιγότερο αποτελεσματική, βλέπει τα πράγματα και τα μελετά λίγο περισσότερο, αλλά δεν είναι πολύ αποδοτική. Και τρίτη, ε, σενάριο καταστροφικό, οικονομική κρίση, άλλα προβλήματα που θα μας οδηγήσουν στο να συνεχίσουμε να εξαρτώμεθα τόσο πολύ από τα καύσιμα τα οποία εισάγουμε κυρίως από τρίτες χώρες. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία μοντέλα που επεξεργαστήκαμε, τα συγκρίναμε, και είπαμε ότι ανάλογα με τους στόχο θέλουμε να υλοποιήσουμε ποια είναι τα μέτρα τα οποία θέλουμε να υιοθετήσουμε. Βεβαίω, το τρίτο σενάριο της καταστροφής δεν το συζητάμε, είναι υποθετικό, είναι θεωρητικό. Και καταλήξαμε στο εξή συμπέρασμα. Αν θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη και αν κατορθώσουμε να έχουμε μια τέτοια ισχυρή Ευρώπη που θα κάνει τι κατάλληλε επενδύσει, αν θέλουμε να υλοποιήσουμε το στόχο αυτό λοιπόν, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη διάφορα στοιχεία τα οποία θα συνδυάσουμε δεδομένου ότι δεν υπάρχει μία λύση αποτελεσματική από μόνη της. Δηλαδή, συνδυασμών, συνδυασμός ε, ε, μορφών ενέργειας που θα χρησιμοποιούμε, συνδυασμός μέσων βάσει των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν, διάφοροι τρόποι χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τεχνολογιών και βεβαίως κίνητρα για να γίνουν επενδύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Κατά την άποψή μου αυτή η άσκηση που θέλετε που έγινε ήταν χρήσιμη. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ούτως ή άλλως αυτά τα θέματα θα συνεχίσουμε να τα συζητούμε ακόμη για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και ο καθένας θα πει ποια είναι η γνώμη του και ποια είναι η απόψή του από πολιτικές πλευράς, αλλά είναι σαφές ότι αν θέλουμε να έχουμε καλής ποιότητας και βιώσιμα ε, δίκτυο μεταφορών στην Ευρώπη θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες. Επίσης, τελειώντας, θέλω να πω ότι ως Επιτροπή Μεταφορών και για το μέλλον θα πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί, πιο δυναμικοί, πιο δραστήριοι. Σε σχέση με αυτά τα οποία μας, μας προσφέρει η ΣΤΟΑ. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρουμε με περισσότερη σαφήνεια τι ακριβώς θέλουμε δεδομένου ότι εκτός από αυτά τα οποία προτείνει υπάρχουν και άλλοι τρόποι τους οποίους μπορούμε να ερευνήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν για την επόμενη θητεία να γίνουν οι κατάλληλες επιλογές και οι σωστές επιλογές γιατί οι μελέτες αυτές ε, θα πρέπει κάπου να καταλήξουν, να μην πάνε. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο ζητάει η συνάδελφος Τικάου. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι πήρα μέρος ε, σε μερικές εκδηλώσεις που οργάνωσε η ΣΤΟΑ που αφορά τις μεταφορές, ενδιαφέρουσες μελέτες. Έχω να κάνω και μία σύσταση. Μέσω της ΣΤΟΑ πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε μελέτες που αφορούν τα έξυπνα συστήματα μεταφοράς. Για το κόστος, πώς θα εσωτερικευτεί, χρειάζονται μελέτες. Βάση για μελλοντικέ συστάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω όντως ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι θα έρθουν στο νέο κοινοβούλιο στο Σεπτέμβριο θα έπρεπε να συνέλθουν σε σώμα και να συζητήσουν τι νέες εκθέσεις θα ζητήσουμε από, το, από τη ΣΤΟΑ. Είναι πολύ καλή δυνατότητα για να έχουμε γενικές πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στην εργασία μας και γι' αυτό ε, θα πρέπει στην πρώτη συνεδρίαση ε, της Επιτροπής ε, Μεταφορών του Σεπτεμβρίου να τεθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη κατά τρόπον ώστε να δούμε ποια είναι τα νέα θέματα τα οποία πρέπει να επεξεργαστούν και η Μπάρση Πατάκη ίσως και άλλοι να αναλάβουν πάλι τις, τα ίδια καθήκοντα διότι τα έχουν καταφέρει πολύ καλά και δεν πρέπει να τους χάσουμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που ζητά τον λόγο, αν όχι τότε θέλω να ευχαριστήσω του τους ε, εκπροσώπους μας ε, στην Επιτροπή στο Α, ε, την κυρία Μπάρση Πατάκη και θα παρακαλούσα όσους δεν είναι συντονιστές να εξέλθουν από την αίθουσα γρήγορα διότι θα κάνουμε αμέσω την συνεδρίαση των συντονιστών εάν εξέλθουν όλοι αυτοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των συνδυαστών. Άρα σε 3,5 λεπτά θα κάνουμε